meine Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσει η συνεδρίαση. Να ξέρω, ίσως συμμαζευτούν και λίγο οι εισηγητές. Αλλά και βέβαια προσπαθώ εδώ και 25 χρόνια και δεν τα καταφέρνω exactly that. <laughs> I never ever, I never ever pay attention to it. <laughs> Ich äh, freue mich, äh, dass. Χαίρομαι για το ότι έχουμε ένα ενδιαφέρον πάνελ στην ε, σημερινή ακρόαση και νομίζω θα έχουμε μια καλή συζήτηση. Είναι πολύ ενδιαφέρον σήμερα το, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση Γερμανίας αποφάσισε να στείλει δύο πυροβολαρχίες ε, Patriot με 400 άτομα προσωπικό στα σύνορα της ε, Τουρκίας ε, για να την προστατεύσει από την Συρία. Ε, και αφενός βεβαίως είναι κάτι αυτονόητο εντός του ΝΑΤΟ και βεβαίως είναι και ενδιαφέρον γιατί στη δημόσια συζήτηση λένε πού μπλέκουμε ξέρουμε πραγματικά ποιοι είναι οι στόχοι της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και δεν ήταν ε, ποτέ πιο εντατική αυτή η συζήτηση από ό,τι σήμερα για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν Ας δούμε τα τυπικά. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι υποψήφια χώρα για τα ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου θα συζητήσουμε. Και τρίτον, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, η Τουρκία σήμερα είναι σημαντικότερη για στρατηγικούς λόγους από ό,τι και στον καιρό του ψυχρού πολέμου. Για τον λόγο αυτό θεωρώ πως ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε συμφέρον για μια σταθερή εξέλιξη της ε, κατάστασης γιατί αν δει κανείς το χάρτη βλέπουμε πως η Τουρκία ως ένα κράτος δικαίου και δημοκρατία και ως μια χώρα η οποία έχει κοινά συμφέροντα και είναι σύμμαχος με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ Νομίζω πως ε, ακολουθεί μια πολιτική θετική. Επίσης ε, έχουν αλλάξει σχέση με το Ισραήλ τα τελευταία δύο χρόνια. Υπάρχει κάποια ασάφεια όσον αφορά τις ε, προσπάθειες διαμεσολάβησης με το Ιράν και τα όχι και τόσο ξεκάθαρα κίνητρα αυτής της πολιτικής η πολιτική την οποία ασκεί ασκούσε η Τουρκία για τους ε, τουρκόφωνους ε, πληθυσμούς ε, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Βεβαίως υπάρχει και η κατάσταση στην Συρία. όλα αυτά. Αυτή η πολιτική λοιπόν απέναντι στη Συρία είναι παρακολούθημα της πολιτικής της Ευρωπαϊκή Ένωσης και του ΝΑΤΟ ή είναι μια πολιτική με την Τουρκία στο επίκεντρο. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν κάποιες ε, ανασφάλειες ε, και αμφιβολίες αλλά ούτως ή άλλως ε, καμιά φορά έχουμε την αίσθηση πως τονίζεται η αυτονομία της Τουρκίας για να πούνε προς ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορούμε και αλλιώς αν θέλουμε ή ότι εκεί υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα ότι η Τουρκία μπορούσε πράγματι να ακολουθήσει έναν άλλο τρόπο. Είναι λοιπόν ε, η Τουρκία ένα κοσμικό κράτος ή υπάρχει η πιθανότητα λόγω της αυξανόμενης Ισλαμοποίησης να υπάρξουν και άλλοι εταίροι. Ε, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σήμερα με τους ε, ειδικού μας. Χαίρομαι εδώ πέρα που έχουμε την κυρία Σένε Μαϊντίν, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μπιλγκή της Κωνσταντινούπολης. Καλώς ήρθατε είναι εδώ πέρα και ο Νιγκάρ Γκιοξέλ, αναλυτής ε, του European Stability Initiative και ο Γκίντερ Ζόιφετ, ο οποίος είναι ε, επιστημονικός ε, συνεργάτης του Πανεπιστημίου Ασφάλειας και Πολιτικής του Βερολίνου αλλά και ο πρέσβης ο κύριος Μωρίς Ριπέρ από την, από την Άγκυρα, ο οποίος ήρθε και θα πρότεινα να ξεκινήσει ο πρέσβης να μας παρουσιάσει την θέση του, μετά θα αναλάβει την Προεδρία ο σύνολος ο κύριος Σορκόβατσεφ. Κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σιγητά, διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί φίλοι. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά που μου δίνετε τη δυνατότητα να απευθυνθώ στην Επιτροπή σας. Πριν στραφώ στην εξωτερική πολιτική, λίγα λόγια αν μου επιτρέπετε για την κατάσταση πραγμάτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Το θίξατε στην εισαγωγή σας. Η έκθεση προόδου για το 2012 που συνετάχθη για το κράτος δικαίου για όλες τις χώρες υποψήφίε προκάλεσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, στην Τουρκία 200 άρθρα στον τύπο δύο εβδομάδες μετά τη δημοσίευσή της και σε μεγάλο βαθμό η μεγάλη πλειονότητα των ε, αντιδράσεων αντίθετα από ό,τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς όλοι λοιπόν ε, το 85% η μεγάλη πλειονότητα με βάση τη μελέτη που κάναμε άρθρα πανεπιστημιακά άρθρα και τέτοια τονίζουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί αλλά και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η περαιτέρω πρόοδος. Η επίσημη τουρκική αντίδραση ήταν επικριτική. Τόνισε ότι ε, τονίζεται υπερβολικά αυτό που πρέπει να γίνει και όχι επαρκώς ότι έχει επιτευχθεί. Έγινε λοιπόν έντονη συζήτηση και νομίζω ότι για το Κοινοβούλιο θα ήθελα να πω κάτι που έχω επανειλημμένα πει. Υποτιμούμε τη σημασία των επιτευγμάτων και ίσως εστιάζουμε κάπως υπερβολικά σε ό,τι απομένει να γίνει. Αν και βέβαια είναι αποστολή μας να αξιοποιούμε τις εκθέσεις προόδου ως οδικούς χάρτες για τα τεκτενόμενα έγιναν σημαντικές αλλαγές φέτος. Όλοι αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας και η επαναβεβαίωση της δέσμευσης της Ένωσης, τουλάχιστον από την Επιτροπή για την ένταξη της Τουρκίας, ε, ήταν σημαντική, αλλά πολλά πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές. Υπήρξε έντονη αντίδραση των αρχών της Τουρκίας, ήταν έκφραση απογοήτευσης γιατί όπως ξέρετε δεν έχει ανοίξει κανένα κεφάλαιο για διαπραγματεύσεις από τα μέσα του 2010. Τα κράτη-μέλη της Ένωσης θεωρούμε ότι φέρουν κάποια ευθύνη. Όπως είπε και ο Επίτροπος Φίλε όταν παρουσίασε την έκθεση στο Κοινοβούλιο. Στην Τουρκία η κατάσταση πραγμάτων της διαδικασίας ένταξης θεωρείται ότι δεν προχωράει διότι υπάρχουν κάποιες διακρίσεις, ε, είναι άδικο το καθεστώς διαπραγματεύσεων για την Τουρκία, διότι υποτίθεται ότι αυξάνεται ο Ισλαμισμός. Επίσης, ε, οι προκλήσεις που δημιουργεί για την Ευρώπη η οικονομική επιτυχία της Τουρκίας και φυσικά το θέμα της Τουρκίας. Είναι σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε πολιτικά την κατάσταση. Είναι σαφέ ότι υπάρχει λιγότερο ενθουσιασμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα, παρά το ότι ίσω. Ε, Δύο θέματα συγχέονται εάν θεωρούν οι Τούρκοι ότι θα ενταχθούν ποτέ στην Ένωση και αν επιθυμούν αυτή την ένταξη. Αλλά ο τρόπος που αντιλαμβάνονται πολιτικά έχει να κάνει με την ουσία των σχέσεων Ένωσης Τουρκίας, αλλά συνολικά από πλευράς εμπορίου ή το 45% της Τουρκίας είναι με τις χώρες της Ένωσης, πολιτιστικές ανταλλαγές, 50.000 ε, φοιτητές και πανεπιστημιακοί και μέλη Ινστιτούτων έρχονται στην Ευρώπη και δαπάνησαν πάνω από 850 εκατομμύρια φέτος. Πρέπει να ενισχύσουμε τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου, να υπάρξει ένα νέο σύνταγμα που θα επιλύσει κάποια μακροχρόνια και περίπλοκα προβλήματα όπως το κουρδικό και που να είναι εναρμονισμένο με τις πρακτικές και τις προσδοκίες της Ένωσης. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να επιτύχουμε το τέταρτο πακέτο δικαστικών διαπραγματεύσεων και επίσης πρέπει να προχωρήσει η συνταγματική διαδικασία που κατά τη γνώμη μου ε, παραμένει ζωντανή παρά τις δυσχέρειες. Ο πρόεδρος Γκουλ παραμένει ισχυρά αφοσιωμένος όπως είπε και την 1η Οκτωβρίου στη διαδικασία ένταξης και πολύ σημαντική είναι η αλλαγή τόνου του Πρωθυπουργού. Πρέπει να υπογραμμιστεί. Όλοι συμφωνούμε με τα σχόλια που έκανε στο Βερολίνο την 1η Νοεμβρίου ότι η Τουρκία και η Ένωση είναι αμοιβαία απαραίτητη για τις οικονομίες των μεν και των δε. Οι Υπουργοί ε, Εσωτερικών, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης εργάζονται και συνεργάζονται και προσπαθούμε να εναρμονίσουμε. Συμφωνώ και με τα σχόλια του Υπουργού Μπαΐς που είπε ότι το κοινό συμφέρον και οι ταχαίως μεταβαλλόμενες παγκόσμιες δυναμικές κάνουν την ένταξη της, Ένωσης, της Τουρκίας στην Ένωση απαραίτητη. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα νέο πολιτικό συμβόλαιο, να επαναζωογονηθούν οι διαπραγματεύσει και να αποκτήσει περισσότερη αξιοπιστία και για μας και για το λαό της Τουρκίας η διαδικασία ένταξης. Να επανέλθει λοιπόν η εμπιστοσύνη. Πέρα από το θετικό θεματολόγιο που όπως ξέρετε επιτυγχάνει αποτελέσματα. Με την επερχόμενη Ιρλανδική Προεδρία προσβλέπουμε στην προσπάθεια καθορισμού ενός οδικού χάρτη για το πρώτο τμήμα του 2013 να συνεχίσουν, να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για τις προξενικές θεωρήσεις, για τον τομέα της ενέργειας, περισσότερες επαφές στην εξωτερική πολιτική κτλ. Εξωτερική πολιτική. Όπως λέει όπως και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσεως, έχουμε επενδύσει πολύ στην ενίσχυση του διαλόγου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την κυρία Άστον. Είναι τμήμα της εντολής που έχει δώσει την υπηρεσία της. Όπως πολλές χώρες, η Ένωση και η Τουρκία θα μπορέσουν να ωφεληθούν από την ε, ενίσχυση της συνεργασίας αυτό θα έχει επιπτώσεις και στα Δυτικά Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή και στην ε, Βόρεια Αφρική και φυσικά και στο Αφγανιστάν και την Νοτιοανατολική Ασία, ολόκληρη την Ασία και σε πολύ στρατηγικό επίπεδο θα βοηθήσει τις σχέσεις μας, τις σχέσεις μας με τον Ισλαμικό κόσμο. Το 2012 η Τουρκία και η Ένωση είναι σε επίπεδο συνεργασίας παρόμοιο και σε ορισμένες περιπτώσεις μεγαλύτερο από κάποιες μεγάλες χώρες. Υπάρχει διάλογος, υπουργικές συναντήσεις, διαβουλεύσεις για το συντονισμό της πολιτικής, επαφές σε επίπεδο ε, διευθυντών πολιτικής των Υπουργείων, διάλογος για την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, τον κόλπο, τα Δυτικά Βαλκάνια. Και φυσικά υπήρξε και μια, διά, μια διάσκεψη που οργανώσαμε μαζί με τα επιμελητήρια στην Κωνσταντινούπολη τον Οκτώβριο για το παγκόσμιο εμπόριο για να υπάρξουν επενδύσεις στην Αίγυπτο, την Τινησία και την Παλαιστίνη. Η Τουρκία υποστηρίζει τις προσπάθειες για το κέρας της Αφρικής και το Σουδάν και θέλει να συμμετάσχει. Συγγνώμη, όχι, της προτάθηκε να συμμετάσχει, αλλά ακόμη δεν έχει απαντήσει. Τώρα δεν έχω πείρα από τη συμμετοχή της Τουρκίας σε επιχειρήσεις μη στρατιωτικού χαρακτήρα, αλλά ίσως από τα κράτη-μέλη εδώ να υπάρχει περισσότερη απροθυμία. Όπου μπορούμε λοιπόν εργαζόμαστε μαζί, εφόσον έχουμε κοινούς συνομιλητές και θεωρούμε ότι από κοινού δράση ενισχύει τη δράση μας. Προσπαθούμε να βασιστούμε στις κοινές μας αξίες αλλά και τις ε, ε, ιδιοτυπίες μας. Μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Υπάρχουν συγκεκριμένες προκλήσεις. Η στάση της Τουρκίας για την συνεργασία με την Κύπρο είναι ένα θέμα που μειώνει την συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Προσπαθούμε να συντονιστούμε με την κοινή πολιτική εξωτερικών και άμυνας και αυτό είναι μια πρόκληση. Αλλά δεν θα πρέπει οι ουσιαστικές συγκλήσεις να ε, συγχέονται με την επίσημη δημόσια ταυτόσιμη αντιμετώπιση. Αλλά να έχετε υπόψη ότι μόνο πρόσφατα η Τουρκία επανακαθόρισε τον ρόλο της στην εξωτερική πολιτική μετά από έτη συζήτησης. Διότι στο παρελθόν είχαμε μια αντιμετώπιση που βασιζόταν σε θέματα ασφάλειας. Άρα ακόμη ανακαλύπτει το χαρακτήρα της εξωτερικής πολιτικής της, αλλά πάντα βέβαια στα πλαίσια της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Η Τουρκία μπορεί να μην έχει ακόμη τα εργαλεία να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες της ή να έχει διαφθρωμένο διάλογο με την Ένωση για τα διάφορα θέματα. Η αναπτυξιακή βοήθεια και η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ουσιώδη στοιχεία της ε, εξωτερικής δράσης της Ένωσης που παραδοσιακά όμως δεν έπαιζαν μεγάλο ρόλο στην τουρκική εξωτερική πολιτική. Τώρα όμως αυξάνεται αυτή η τουρκική πολιτική, πρόκειται για δισεκατομμύρια, αλλά το εμπόριο και οι επενδύσεις μπορούν να βοηθήσουν, γιατί για παράδειγμα αυξάνεται η τέτοια οικονομική παρουσία της ε, Τουρκίας στην Αφρική. Επίσης μπορούμε να αξιοποιήσουμε το δίκτυο των μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν χτίσει σχολεία σε διάφορα μέρη της Ασίας και της Αφρικής. Ή ιδρύματα. Σε πολλές περιπτώσεις η Τουρκία μοιάζει να μην συνδυάζεται με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θεωρεί ότι οι δυτικέ πρώην επικιακές δυνάμεις δεν είναι ο πιο κατάλληλος φορέας. Ενώ η τουρκική προσέγγιση, δηλαδή Ισλάμ συνδημοκρατία... δημοκρατία, θεωρεί η Τουρκία ότι είναι ελκυστική για ε, πολλές χώρες. Αυτός είναι για παράδειγμα ο τρόπος με τον οποίο προωθούμε την πολιτική μας στην Αφρική, ιδίως στη Σομαλία. Παρά τις προσπάθειες λοιπόν του κυρίου Ταβούτογλου και παρά τους ε, φιλόδοξους στόχους που έχουν προκηρυχθεί για τη Μέση Ανατολή και τα Δυτικά Βαλκάνια και άλλες περιοχές, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας δεν μας δίνει ακόμη μια 100% σαφή εικόνα για τις προθέσεις και τα αποτελέσματα. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι η τουρκική πλευρά θέλει να συνεργαστεί με την Ένωση για την κρίση στη Συρία. Η Τουρκία είναι στην πρώτη γραμμή και η πρόκληση είναι η Τουρκία να αποτρέψει περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας στη Συρία, να σταματήσει τη μαζική εισρωή προσφύγων. Αυτή τη στιγμή Έχουμε σε στρατόπεδα 130.000 άτομα σε στρατόπεδα και 70 με 100.000 περαιτέρω στη χώρα και ίσως και πάνω από 20.000 στα σύνορα. Τελευταίο, τελευταίο στόχος της Τουρκίας είναι να υπάρξει μια επιτυχής και ταχεία μετάβαση στη Συρία. Εφόσον μιλάμε για την τουρκική θέση έναντι της Συρίας, ένας από τους βασικούς στόχους εξωτερικής πολιτικής είναι να αντιμετωπιστεί και το κουρδικό ζήτημα. Θέλουμε να προωθήσουμε μία ε, συμμαχία αντικυβερνητική χωρίς αποκλεισμούς στη Συρία για να μην υπάρξουν επιπτώσεις ε, της κρίσης αυτής για την Τουρκία εάν υπάρξει μία περίπου ανεξάρτητη αυτόνομη κουρδική περιοχή στη Βόρεια Συρία όπως το Ιράκ. Βλέπουμε ότι συγκλίνουμε για τη Βόρεια Αφρική. Βοηθάμε τις αναδυόμενες δημοκρατίες και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια τρομοκρατία. Η Τουρκία από το 2011 είναι συμπρόεδρος του Παγκόσμιου Φόρουμ κατά της τρομοκρατίας στην Αφρικα και την Ιεμένη. Στη διαδικασία ειρήνευσης της Μέσης Ανατολής η Τουρκία ήταν στο προσκήνιο της ε, πάλης για την αναγνώριση της Παλαιστίνης και εξακολουθούμε να ε, Είμαστε αντιμέτωποι με το κράτος του Ισραήλ. Οπωσδήποτε η επιδείνωση των σχέσεων Τουρκίας-Ισραήλ, της Συρίας, του Ιράκ και του Ιράν δεν βοηθάει την Τουρκία για να παίξει κεντρικό ρόλο στην Μέση Ανατολή. Η πυρηνική κρίση με το Ιράν είναι άλλη μια ευκαιρία για διάλογο Ένωσης και Τουρκίας. Κάποια στιγμή η Τουρκία εξέφρασε την επιθυμία να ενταχθεί σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Υποστηρίζουμε την δυτή προσέγγιση και είμαστε πάντα διατεθειμένοι να περάσουμε μηνύματα αμφίδρομα. Ιδίω γιατί οι πιο πρόσφατες συναντήσει έγιναν στην Κωνσταντινούπολη. Η Τουρκία έχει απτά αποτελέσματα σε τριμερή διάλογο με το Πακιστάν και το Αφγανιστάν διότι η Τουρκία, όπως ξέρετε, φιλοξένησε στην Κωνσταντινούπολη τον περασμένο Νοέμβριο μια τριμερή συνάντηση κορυφή και την διεθνή διάσκεψη για το Αφγανιστάν και επίσης στην Άγκυρα έγινε τον Οκτώβριο η συνάντηση της ομάδας επαφής για το Αφγανιστάν. Η Τουρκία παίζει αυξανόμενο ρόλο σε πολυμερή φόρα. Είμαστε στο ΝΑΤΟ και τον ΟΣΑ αλλά και σε άλλους φορείς. Ο Ερντοάν πήγε στο Πακιστάν πρόσφατα για να ε, παραστεί στη συνάντηση κορυφή του D8 και στο G20 το 2015. Θα προσπαθήσουμε να επανεκλεγούμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επίσης σημειώνουμε ότι στην Τουρκία είναι η γραμματεία του Μπισεκ και είμαστε και ε, πρόεδροι της οργάνωσης του της Ισλαμικής οργάνωσης. Η Τουρκία επίσης είναι η 16η οικονομία του πλανήτη σήμερα. Προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή της, να αναλάβει περισσότερες ευθύνες στην λήψη αποφάσεων στον πολιτικό τομέα. Οι επιπτώσεις της τουρκικής προσπάθειας δεν είναι ακόμη πολύ σαφείς, διότι η εξωτερική μας πολιτική δεν έχει αρκετή πείρα και για την ε, παγκόσμια οικονομική κατάσταση και για την ε, συζήτηση για την αλλαγή του κλίματος, την ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις, προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού, θέλουμε να αφοσιώσουμε περισσότερες προσπάθειες. Οι απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις, κατά τη γνώμη μου, είναι πιο επίσημος διάλογος, περισσότερες διαβουλεύσεις με την Τουρκία και σε επίπεδο ε, Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία screening του κεφαλαίου 31 για το κεκτημένο που ελπίζουμε να επιτύχουμε μέχρι τον Ιανουάριο του 2013. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη για την εισαγωγή αυτή. Προτείνω τώρα να ακούσουμε τους ειδικού μας και μετά βεβαίως και την εισηγήτρια. Θα ήθελα Πρώτα απ' όλα λοιπόν να δώσω τον λόγο στην κυρία Τζγκίτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρέσβη για την εισαγωγή αυτή. Η δική μου η παρέμβαση λοιπόν θα κινηθεί κυρίως στο πλαίσιο του ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και η προβληματική τομή της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να τονίσω πως εάν θέλουμε να καταλάβουμε την τουρκική εξωτερική πολιτική πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά τις ε, εξελίξεις στο ιστορικό της Τουρκίας γιατί συνδέεται η γραμμή του ΑΚΠ στα εξωτερικά με την εσωτερική πολιτική και τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Τουρκίας. Όταν προσπαθεί κανείς να αναλύσει τις εξελίξεις ε, μπορεί να σε τέτοιο πλαίσιο μπορεί να εξηγήσει την πολιτική και το προσανατολισμό του ΑΚΑΠΕ που αυτή τη στιγμή βεβαίως ε, κινείται πιο πολύ προς την κατεύθυνση πρωτοβουλειών που θεωρείται πως θα τα εκτιμήσει ο τουρκικός λαός ε, για να προωθήσει τον Ερντογάν στην ε, Προεδρία. Πρέπει να τα έχουμε αυτά κατά νου. Γιατί βεβαίω υπάρχουν και στην συζήτηση στο εσωτερικό της Τουρκία. Και βεβαίω αυτό υπονοεί πως ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή ε, κυρίως ε, ασχολείται με το εθνικό, εθνικιστικό σώμα, με αυτούς τους ε, του. Γι' αυτό κάνει συχνές αναφορές ε, στη λεγόμενη Οθωμανική κληρονομιά, στους προγόνους μας, ε, και στον τουρκικό ακτιβισμό στην ευρύτερη γειτονιά μας και νομίζω πως εξηγεί και την μεταστροφή και στο κουρδικό. Όλα αυτά νομίζω μπορούν να ερμηνευθούν ως μέρος ενός πακέτου που έχει σχέση με την εσωτερική πολιτική και με την πιθανότητα δημοψηφίσματος για ένα πιο προεδρικό σύστημα στην Τουρκία, το οποίο θα ήθελε ο Ερντογάν. Έχοντας θέσει αυτό ως πλαίσιο λοιπόν, νομίζω πως τώρα μπορούμε να εστιαστούμε σε δύο τομείς για να συζητήσουμε την τουρκική εξωτερική πολιτική. Ο ένας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ζήτημα εξωτερικής αλλά και εσωτερικής πολιτικής και βεβαίως ε, τη Μέση Ανατολή. Όταν λοιπόν ε, ξεκινάμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλεγα πως όλοι μπορούμε να πούμε πως οι σχέσεις μας ε, έχουν ε, μία στασιμότητα. Βεβαίως αφενός βλέπουμε πως υπάρχει κάποια πρόοδος παρά το ότι δεν μπορούν να κλείσουν οι διαπραγματεύσεις και τα κεφάλαια. Υπάρχει μια τεχνική ευθυγράμμιση πολλή δουλειά η οποία γίνεται στα Υπουργεία, οπότε στο τεχνικό επίπεδο υπάρχει πρόοδος, αλλά κανείς δεν τα αναφέρει αυτά γιατί υπάρχει στάσιμότητα στην ε, πολιτική σχέση των δύο πλευρών. Και αυτό είναι ανησυχητικό αφενός για, το, για τις συνέπειες που έχει, αλλά από την άλλη βεβαίως δείχνει πως ε, όταν ξεπεραστούν τα πολιτικά εμπόδια υπάρχει ήδη ένα μεγάλο, αρκετά μεγάλο ποσοστό ευθυγράμμισης. Βεβαίως, υπάρχουν, ε, υπάρχει και αντίκτυπο στην εσωτερική πολιτική της Τουρκίας. Πρώτα απ' όλα αυτό σημαίνει πως ε, συνεισέφερε, χωρίς να είναι ο μόνος ε, παράγων, στην στασιμότητα της, του δημοκρατικού μετασχηματισμού της Τουρκίας. Και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Και αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους. Αφενός ε, υπήρχε η μειωμένη αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και βεβαίως αυτό σήμαινε πως ε, έχει μειωθεί και η στήριξη του κοινού για την ένταξη της Τουρκίας. Και βεβαίως υπάρχει και εσωτερική πτυχή αυτής της συζήτησης γιατί υπάρχει το ζήτημα αυτού που εγώ αποκαλώ την ε, διαφοροποίηση όσον αφορά την αυτονομία της τουρκικής ελίτ. Δηλαδή χρησιμοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση από την κυβέρνηση για να αποκτήσει μια κάποια νομιμότητα στα μάτια των πιο κοσμικών, της γραφειοκρατίας, της διοίκησης κτλ. Τώρα αυτή η ανάγκη φαίνεται πως ε, δεν ισχύει τόσο πολύ οπότε η ρεαλιστική βάση για, την, ε, για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της κυβέρνησης φαίνεται πως επίσης δεν υφίσταται. Οπότε μαζί με τα αντιφατικά μηνύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προοπτική ένταξη της Τουρκίας δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο όσον αφορά τις πολιτικές ε, μεταρρυθμίσεις και έχει αυτό βεβαίω συνέπειε και για την εξωτερική πολιτική της, ε, στι οποίε θα επανέλθω. Τι είναι η πτυχή λοιπόν ε, των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για τη Μέση Ανατολή, όπως είπε και ο κύριος ε, Πρέσβης, έχουμε δει μια Τουρκία η οποία δρά χωρίς να αντιδρά απλώς στα γεγονότα. Έχουμε την περίφημη πολιτική μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες που πήγε καλά μέχρι το 2011 και το 2011 ήταν ένα έτος κρίσιμο. Ε, σε δύο ε, μέτωπα. Δηλαδή αφενός ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη και κάτι που είναι εξίσου σημαντικό και δεν αναφέρεται συχνά είναι πως ε, τότε έφυγαν οι Ηνωμένε Πολιτείε από την περιοχή και αυτό έχει ουσιαστική σημασία όσον αφορά την αλλαγή ισορροπιών στην ε, περιοχή. Οπότε αυτές οι δύο ε, εξελίξεις άλλαξαν το πεδίο. Μέχρι τότε ήταν αρκετά επιτυχής η εξωτερική πολιτική, δηλαδή υπό την έννοια πως βεβαίως υπήρχαν προβλήματα αλλά υπήρχαν συγκεκριμένα αποτελέσματα όπως η προσέγγιση με τη Συρία, διευκόλυνση βίζας ε, και απελευθέρωση με πολλές χώρες ε, της περιοχής, Συρία, Λίβανος, ε, Ιεμένη κτλ. Και βεβαίως αυξημένη οικονομική αλληλεξάρτηση, διασυνοριακό εμπόριο. Οπότε οικονομικά και πολιτικά ήταν ε, μια εποχή επιτυχημένης ε, τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Η Τουρκία ακολουθούσε μια πολιτική και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με μια πιο περιφερειακή έμφαση που υλοποιήθηκε σε πολλούς τομείς στην περιοχή. Κάτι το ενδιαφέρον βεβαίως είναι πως πριν το 2011 και την Αραβική Άνοιξη η πολιτική αυτή δεν είχε κάποια αιρεσιμότητα. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι το αντίθετο με την ε, ευρωπαϊκή πολιτική. Όταν λέω αυτό τι εννοώ. Και βέβαια αυτό ήταν ε, και κάτι για το οποίο ήταν υπερήφανη η Τουρκία. Δηλαδή η δημοκρατία και η πρόθεση δημοκρατίας δεν ήταν σημαντικό ζήτημα. Οπότε βεβαίως μόλις δεν ασχολείται κανείς με αυτό ήταν ε, εύκολο να έρθει σε επαφή με κάποια από τα προηγούμενα καθιστώτα στην περιοχή. Οπότε ήταν ζήτημα οικονομικών σχέσεων και όχι απαιτήσεων. Και υπήρχε πάντα βεβαίως και αυτό το οποίο ε, υπονοούσαμε πως αν δεν μας στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουμε και άλλες επιλογές και νομίζω πως αυξήθηκε έτσι και η δημοτικότητα και της Τουρκίας και του Ερντογάν θα έλεγα προσωπικά και έλεγαν διάφοροι πως η ήπια ισχύση της Τουρκίας αυξάνεται κτλ. Βεβαίω μετά την Αραβική Άνοιξη και το 2011 τα πράγματα αλλάζουν. Βεβαίω είδαμε πως η πολιτική αυτή ε, τις μη, χωρίς όρους ε, για τη δημοκρατία, δεν έστεκε η δε πολιτική μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες, δεν μπορούσε να ακολουθεί οπότε έπρεπε να αλλάξει. Και έγινε αυτό. Προσαρμόστηκαν με το να συνταχθούν με τις δυνάμεις αντιπολίτευσης ε, και γρήγορα, αλλά και εκεί πέρα υπήρχαν προβλήματα, παραδείγματος χάρη ε, στην Συρία, που εγώ προσωπικά δεν βλέπω ως προέκταση της Αραβικής Άνοιξης αλλά μια κατάσταση σαν το Λίβανο του 1970 έναν εμφύλιο πόλεμο και μια περιφερειακή σύγκρουση δηλαδή έρχονται και άλλοι παράγοντες εκεί. Βεβαίως ετέθη και το ζήτημα των επαφών με τους αδελφούς ε, μουσουλμάνους και υποτιμήθηκε βεβαίως ε, και η ισχύ ε, του καθεστώτος που έχει κάποια στηρίγματα στην ε, κοινωνία και ειδικά η Συρία έδειξε γιατί το ΑΚΠ ε, παραδοσιακά ασκούσε κριτική και μαλιστές ότι δεν καταλαβαίνουν την περιοχή, αγνοούν την περιοχή αλλά αυτό έχει δείξει πως και το κυβερνών κόμμα δεν ε, αντιλήφθηκε πλήρως την περιοχή και υπερτιμούσε την γνώση της περιοχής και του ρόλου που μπορεί να παίξει η Τουρκία. Ε, αυτό το οποίο συνέβη μετά την Αραβική Άνοιξη είναι πως ε, όλα αυτά τα οποία λέγαν για τουρκικό μοντέλο κατέληξαν να αφορούν το μοντέλο του ΑΚΑΠΕ. Δηλαδή το εάν οι νέοι Ισλαμιστές ε, θα έκαναν έναν εκδημοκρατισμό τύπου ΑΚΑΠΕ. Και βεβαίως έδειξε και τα όρια του μοντέλου αυτού γιατί αποξένωσε τις μη Ισλαμιστικές δυνάμεις οδήγησε την Τουρκία στο να κατηγορηθεί για στενούς δεσμούς με τους αδελφούς μουσουλμάνους και βεβαίω υπήρχαν ε, και τα όρια της δημοκρατίας Τουρκίας. Δηλαδή μπορούμε να πούμε πως η Τουρκία είναι μια δημοκρατία αν τη θεωρήσουμε μια δημοκρατία εν εξελίξη ακόμα. Η ίδια η τουρκική δημοκρατία έχει τελματωθεί. Και πάλι βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα αξιών και συμφερόντων στην τουρκική εξωτερική πολιτική. Το είδαμε στη Λιβύη, στη Συρία. Είχαμε οικονομικές σχέσεις οι οποίες ε, διακόπηκαν. Είχαμε τους πρόσφυγες. Εδώ τα νούμερα είναι πάνω από 100.000 ε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κράτους. Ε, δημιούργησε ένα περιβάλλον στο οποίο το ΠΚΚ βρήκε στηρίγματα, πράγματα τα οποία ίσως ε, δεν θα είχαν συμβεί. Γιατί αν προσπαθεί κάποιος να γίνει ισχυρός παίκτης στην περιοχή, μετά πρέπει να προσέχει και το μαλακό του, όπως λένε, υποκάστριο. Συμπερασματικά λοιπόν, Πολλέ φιλοδοξέ ιδέε συζητήθηκαν σε σχέση με το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούσε να συνεργαστεί με την Τουρκία και ο κύριο Πρέσβης ανέφερε κάποιου τομεί και μάλιστα υπάρχουν τέτοια ζητήματα όπως παραδείγματο χάρη η Ένωση τη πολιτική Βοήθειας ε, δεσμοί μεταξύ των αντιπροσωπείων, αλλά τίποτα ουσιαστικό. Αυτό το οποίο κάνει η Τουρκία είναι πως συνεργάζεται με μεμονωμένες χώρες και εμένα μου φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει την σημασία της για την κυβέρνηση. Κάτι το οποίο εγώ, το οποίο εγώ βλέπω ε, ως σοβαρό πρόβλημα προς ανατολισμού της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής αλλά και για την ε, μοίρα της ε, δημοκρατίας εντό Τουρκία, γιατί και ο ακτιβισμός στη Μέση Ανατολή νομίζω δεν μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση του θέματος. Ο επόμενος κυρία Μουτσέλα, αναλήτρια Σας ευχαριστώ. Έχω ένα πλεονέκτημα. Συμφωνώ με τόσα πολλά από τα σημεία που αναφέρθηκαν ήδη και αυτό που θα πρέπει να κάνω είναι να οικοδομήσω σε αυτά που ακούστηκαν προκειμένου να μην τα επαναλάβω. Αυτό που προτιθόμουν να πράξω σήμερα είναι ε, τα πόσο η Τουρκία είναι ένα μοντέλο για την μετάβαση στην ε, Μέση Ανατολή και κατά πόσο μπορεί να συμβάλλει ώστε να προωθήσει το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στην ε, περιοχή της, όπως και η δόκτωρ Γκιούζιτς. Θα ήθελα να εξετάζω το θέμα από δύο πτυχές. Ε, μία θα είναι η εσωτερική και η άλλη θα αφορά την δράση της Τουρκίας στην γειτονική περιοχή. Έγιναν σημαντικές αλλαγές τις προηγούμενες δεκαετίες στην Τουρκία έγιναν κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, κοινωνικές αλλογές, κοινωνιακή πρόοδο κλπ. Ε, ακολούθησαν τα δυτικά μοντέλα και φυσικά η ελκυστικότητα της Τουρκίας στην γειτονιά της αυξήθηκε. Τα διδάγματα λοιπόν από τις εξελίξεις στην Τουρκία μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο για τις χώρες της ε, Μέση Θα προσπαθήσω λοιπόν να αναφέρω δύο σημεία και να εκφράσω κάποιες επιφυλάξεις. Εάν ο εκδημοκρατικός της Τουρκίας δεν προχωρήσει ε, μέσω συζητήσεων θα μπορούσε να κατα... έχει αντιπαραγωγικές εξελίξεις και επιρροές και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα εκ νέου του εκδημοκρατισμού. Κάτι ακόμα, ενώ η Τουρκία έχει κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να επηρεάσει το Μέση Ανατολή θετικά, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι κάτι τέτοιο θα γίνει με τον καταλληλότερο τρόπο. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να δυναμωτήσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την ε, στασιμότητα στο οποίο βρίσκεται η κοινωνία της ε, Τουρκίας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει πρωτοβουλία στην περιοχή, ειδικά σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές εξελίξεις, αλλά και τη συμπερίληψη μη κρατικών οργάνων και δομών στην όλη συζήτηση. την περαιτέρω ενίσχυση λοιπόν της κοινωνίας των πολιτών μερικά σχόλια για την εσωτερική διάσταση ενώ τα διδάγματα είναι σημαντικά είναι δύσκολο να μιλήσουμε για το ποιο είναι το μοντέλο Κοιτάζοντα τώρα την Τουρκία όλα τίθενται ένα αμφιβόλο κατά κάποιο τρόπο ποιος είναι ο ρόλος τη θρησκείας τις δικαστικές μεταρρυθμίσεις ε, τις οποίες ενέπνευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και επηρέασαν φυσικά τις ισορροπίες. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι έθεσε το ζήτημα της ε, επανεισαγωγής θανατικής ε, ποινής, θανατικής καταδίκης ε, στην Τουρκία. Ελευθερία έκφραση, ελευθερία του τύπου αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, ορισμένοι δημοσιογράφοι φυλακίστηκαν και είναι δύσκολο λοιπόν να μεταβούν οι Τούρκοι υπουργοί στην περιοχή και να συζητάνε αυτά τα ζητήματα. σε συζήτηση η οποία αφορούσε τα ανθρώπινα δικαιώματα είπαν ότι τα πράγματα, οι Τούρκοι υπουργοί ισχυρίστηκαν ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και η απάντηση ήταν ότι μην μου λέτε αστεία. Οπότε δύσκολα μπορούν να μιλήσουν για πρόοδο και για ένα μοντέλο τουρκικό. Νομίζω πως ε, τώρα έχουν, ε, ε, έχει επιδεινωθεί η κατάσταση στην ελευθερία έκφραση στην Τουρκία. Και πολύ διανοούμενοι κατέληξαν στα δικαστήρια για λόγους ελευθερίας ε, σκέψης και έκφρασης. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση, η κατάσταση μπορούσε να αφορά περισσότερο κράτη-μέλη, τα, κράτη τα οποία δεν ε, προσβλέπουν σε ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, η Τουρκία και η Μέση Ανατολή. Όταν το τηλεοπτικό μοντέλο αναφέρεται, πρόκειται, συνήθως είναι ένα μοντέλο το οποίο αφορά την ε, κόμμα ΑΚΠ. το ΑΚΠ έχει σίγουρα ε, κάποιες επιτυχίες σε ό,τι αφορά την πρόοδο στην Τουρκία. Πολλές φορές όμως, ε, όταν μιλάμε για μοντέλο, είναι δύσκολο να προτείνουμε το τουρκικό μοντέλο σε αφορά τον εκμοκρατισμό. Τώρα, η ε, θέμα της κοινωνίας των πολιτών, ε, η οποία είναι δραστήρια εδώ και αρκετό καιρό, αλλά αυτό ε, αποδόθηκε στο ότι θέλησαν να δώσουν ένα είδος ε, ασυλίας, θα λέγαμε, στην, στον στρατιωτικό τομέα και το φυσικό μοντέλο νομίζω δεν μπορούμε να αποτελέσει πηγή έμπνευση για την περιοχή. Και κάτι ακόμα, παρά τι θετικέ ε, εξελίξει ε, αν δούμε τα αποτελέσματα, νομίζω ότι είναι ανάμεικτα. Οι κυβερνητικοί λένε ότι 2011 στην ε, Αίγυπτο. Αυτά που έγινε στην Αίγυπτο δείχνουν ότι μπορεί να έχετε ένα κοσμικό κράτος, αλλά ε, να υπάρχουν ε, θρησκευτικοί νόμοι που να διέπουν αυτό το κράτος. Η Τουρκία όμως δεν είχε συμμετάσχει στην όλη διαδικασία του φορά το Σύνταγμα της Αιγύπτου. Οι ψηφίες των φιλελευθέρων οι οποίοι ε, διαμαρτύρονταν για την ε, σύνταξη του κειμένου και κατά κάποιο τρόπο λοιπόν ε, η συμμετοχή των νομικών, των διαφωνούντων, των δημοσιογράφων στην Τουρκία αλλά και στην Μέση Ανατολή γενικότερα σίγουρα οδήγησαν σε κάποια απελευθέρωση, αν δούμε ειδικά τα δικαιώματα των γυναικών τα οποία επηρεάστηκαν φυσικά από τα δυτικά συστήματα. Οι χαράσοντες πολιτικοί μίλησαν για σημαντική πρόοδο και για νομικές αλλαγές. Η εμπειρία τους μπορεί να είναι σίγουρα σημαντική για τους Αιγύπτιους, για τις Αιγύπτες μάλλον, για τις τινήσιες γυναίκες και εκλαμβάνοντε ε, τι αποφάσει σχετικά με τι αλλαγέ που απαιτούνται. Το 1999 οι γυναίκε στην Τουρκία χρησιμοποίησαν το μοντέλο τη Μαλαισία. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, όπω καταλαβαίνετε, δημιούργησαν τι ε, εξελίξει, προκάλεσαν τι εξελίξει στην ε, περιοχή. Τώρα, η τουρκική κυβέρνηση έχει επαφές με κάποιους ηγέτες της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον η επιρροή είναι θετική. Μερικές φορές ε, βλέπω ότι οι ισχυρές σχέσεις μεταξύ των ηγετών είναι ένα χάντικα, ένα μειονέκτημα για τους πολιτικούς στην Τουρκία. Όταν βλέπουμε τις σχέσεις των, ε, της Τουρκίας ε, με το Αζερβαϊτζάν ή με τους αδελφούς μουσουλμάνους, οι οποίοι επικρίνουν τις ηγέτες της χώρας, ε, καταλαβαίνετε ότι έχουν αρνητική επίπτωση, επιρροή. Δεν είμαι βέβαιο λοιπόν πως η τουρκική κυβέρνηση είναι το μοναδικό κανάλι μέσω του οποίου ε, ο δημοκρατισμός της Τουρκία θα πρέπει να προχωρήσει. Τελειώνει ο χρόνος μου, θέλω να πω μερικά πράγματα ακόμα. Τώρα τα οι που έχουν γίνει για τον ρόλο της Τουρκίας ε, δείχνουν ότι και ο ρόλος της Τουρκίας ε, έχει κάπως ε, παρεξηγηθεί. Ορισμένοι από τους απαντώντες είπαν ότι οι σχέσεις με, της Τουρκίας με την Δύση αποτελούν ένα μειονέκτημα. Άλλοι από τους ερωτηθέντες είπαν ότι μάλλον είχα ε, ε, άποψη διαφορετική αν η Μέση Ανατολή και ο αραβικός κόσμος ε, είναι ένα στοιχείο το οποίο ενδιαφέρει την Τουρκία, θα πρέπει αυτή η δημοσκόπηση, αυτό η μέτρηση να ληφθεί σοβαρότερα υπόψη. Τώρα, για το θέμα της ε, Ευρώπης θα έλεγα ότι θέτει στο περιθώριο πολλές, πολλούς, ε, πολλά κόμματα στην ε, Τουρκία. και η παρουσίαση του ΑΚΠ ως μοντέλο, ως πρότυπο ε, ε, προβλέπει, μάλλον θεωρείται ως ε, εναλλακτική λύση και υπάρχουν πολλά περισσότερα δίκτυα αλληλεγγύης με την περιοχή και τα εναλλακτικά τμήματα της τουρκικής κοινωνίας έχουν αποδυναμωθεί τόσο στο ιστορικό Τουρκίας όσο και στην περιοχή. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει τα κατάλληλα μέσα για να στηρίξει τον δημοκρατισμό της ε, Τουρκίας Χρειάζεται λοιπόν ένας πιο διαθρωμένος διάλογος με την τουρκική κοινωνία και δεύτερον να ε, εμπλακεί η κοινωνία των πολιτών της Τουρκίας ε, περισσότερο στην διάλογο με τις γειτονικέ χώρε. από όπου έχουν αποκλειστεί πάρα πολλές μη κυβερνικές οργανώσεις. Ευχαριστώ. Και τώρα ο τελευταίος ε, ομιλητής μας, ο κύριος Γκούντερ Σέφερτ είναι συνεργάτης του Γερμανικού Ινστιτούτου για ε, Διεθνείς Υποθέσεις και θα μας μιλήσει για τις αλλαγές στην κοινωνία και την αλλαγή της στρατηγικής ε, επειδή η Γερμανοί είναι πολύ ε, ε, τον παρακαλώ να μιλήσει μόνο 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Όλοι βασιζόμαστε στις προηγούμενες ομιλίες και οι δύο κυρίες αναφέρθηκαν προηγουμένως στις εσωτερικές εξελίξεις πόσο σημαντικές είναι για την εξωτερική πολιτική. Και εγώ προσπαθώ να συνδέσω τις αλλαγές στην κοινωνία και τη νέα βάση της ε, τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Αλλά προσπαθώ να το συνδέσω και με την ε, τωρινή συγκυρία των σχέσεων Τουρκίας μέσα Ανατολής. Ο πρόεδρος κύριος Μπροκ ρώτησε αν η Τουρκία ακολουθεί τη δική της πολιτική ή αν εξαρτάται από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Νομίζω ότι μέχρι πριν από 1,5 χρόνο η Τουρκία είχε δική της πολιτική. Αλλά τώρα και πάλι εξαρτάται από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Θα ήθελα να ε, θέσω το ερώτημα αν θα πρέπει να μας ε, χαροποιεί ή να μας ανησυχεί αυτή η εξέλιξη. Μέχρι πριν από 1,5 χρόνο λέγαμε πολλά για τον ε, ρόλο της Τουρκίας, την ήπια δύναμη, ελεύθερη διακίνηση ατόμων, ιδεών, πολιτιστικών προϊόντων, εμπόριο, ε, η αντιμετώπιση ήταν κοινού συμφέροντος ε, λόγω κοινού πολιτισμού. Βλέπαμε λοιπόν ότι η διπλωματία στην ε, Μέση Ανατολή ξεπέρναγε τις διαφορές. Προσπαθούσαν να δημιουργήσουν περιφερειακές λύσεις σε περιφερειακά προβλήματα. Το είδαμε στον πόλεμο του Ιράκ, στο θέμα του Ιράν, της Συρίας και της Λιβύης. Όλα αυτά ήταν τμήμα μιας προσπάθειας να υπάρξει μια οικονομικά και μετέπειτα πολιτική ενότητα στη Μέση Ανατολή. Αυτό επαναλάμβανε κάποια στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτικής που οδήγησε στη δημιουργία των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Το πιο γνωστό παράδειγμα ήταν η ομιλία του Ερντογάν για το Σέγγεν. Δηλαδή να δημιουργηθεί μια περιοχή χωρίς βίζες. Και ο Τσάι Αγγίλ Υπουργό Εμπορίου, αναφέρθηκε στην ε, ζώνη ευημερία ε, που ήθελε να δημιουργήσει η Τουρκία μαζί με τη Συρία, το Λίβανο κτλ. Αυτή η νέα εξωτερική πολιτική όμως ήρθε σε αντίθεση με τις προσδοκίες ε, των ΗΠΑ και της Ένωσης ιδιαίτερα όσον αφορά την Συρία, το Ιράν αλλά και τη Ρωσία. Και άρα τέθηκε το θέμα ποιος στέει που απομακρύνθηκε η Τουρκία. Παρά όλες αυτές τις κριτικές, η πολιτική αυτή σε μεγάλο βαθμό συνέβαλε στη σταθερότητα και την, ευρωπαϊκή, και την περιφερειακή ενοποίηση. Αλλά βέβαια αυτό μείωσε την άμεση επιρροή Ένωσης είπα. Τώρα και πάλι η Τουρκία επανήλθε στη Δύση λέγεται. Έχει τα ραντάρ κατά της Τεχεράνης, είναι κατά της Ρωσίας στα θέματα της Συρίας. Αλλά η Τουρκία μοιάζει τώρα ε, σχετικά απομονωμένη από τους ε, γείτονές της. Είναι πιο ευάλωτη στο ΠΚΚ και έχει μειωθεί ο ρόλος ηγέτης στην περιοχή. Δεν είναι σε θέση να ε, γεφυρώσει τις διαφορές στην περιοχή. Δεν έχει την ευρύτερη εξωτερική πολιτική που πρόσφατα είχε. Δεν είναι πλέον σε θέση να βοηθήσει την ενοποίηση και την σταθερότητα της περιοχής. Υπάρχει στρατιωτικοποίηση της Τουρκίας πρόσφατα και σε σχέση με τη Συρία και σε σχέση με την Κύπρο. Δεν νομίζω πως αυτό είναι προς το συμφέρον της Ένωσης. Είναι ασταθής η κατάσταση. Από τη μία θα ήταν σκόπιμο να έχει τη δική της εξωτερική πολιτική για να παίξει ρόλο σταθεροποιητή. Και δεν θέλουμε την Τουρκία ναι με να είναι πιο στενά συνδεδεμένη με, την, ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά στην ουσία αναπαράγει τους διαχωρισμούς στη Μέση Ανατολή. Γιατί προέκυψαν όλα αυτά, πώς προέκυψαν. Γιατί δεν μπόρεσε να συνεχίσει την προηγούμενη πολιτική της. Αυτό συνδέεται στενά με εσωτερικές εξελίξεις. Οι κυρίαρχοι πολιτικοί κύκλοι στην Τουρκία θεωρούν ότι ολοκληρώθηκε η εσωτερική πολιτική μεταρρύθμιση, μεταμόρφωση που δημιούργησε νέες προϋποθέσεις για την θέση της Τουρκίας στην περιοχή και για το εσωτερικό της Τουρκίας. Και το κέντρο αυτής της μεταρρύθμισης είναι ένα είδος εκδημοκρατισμού που προέκυψε πρώτον και κυρίως με την ένταξη του μεγάλου συντηρητικού τμήματος του πληθυσμού στην πολιτική και την εκπαίδευση και την οικονομία. Δημιουργήθηκαν νέες πολιτικές και ακαδημαϊκές ελίτ και λειτουργούν και οικονομικές. Αυτές οι νέες μορφές επέτρεψαν στην Τουρκία να αντιμετωπίσει τον ιδιαίτερα ακραίο Ισλαμισμό που ήταν μεγάλη πρόκληση. Ο δυναμισμός των ε, ε, θρήσκων οικονομικών παραγόντων της Ανατολίας βοηθάει την κατάκτηση νέων αγορών και σταματάει λοιπόν όλη αυτή η επιχειρηματολογία ότι οι Ισλαμικές κοινωνίες δεν μπορούν να είναι οικονομικά επιτυχημένες. Και στην εκπαίδευση άλυξε η κατάσταση που παράγει μια νέα συντηρητική οικονομική ελίτ που μπορεί να αναλάβει ηγετικέ θέσει στα πανεπιστήμια, το δικαστικό σώμα, την κοινωνία, τη δημόσια διοίκηση, δημιουργεί μια διαφορετική εκδοχή του τουρκικού κράτους. Βασικά ε, θεμελιώδη δόγματα της μη θρησκευτικής ε, κρατικής δομής τίθενται να αμφιβόλο, δηλαδή η παρέμβαση του στρατού στην πολιτική, η άρνηση της εθνικής πολυμορφίας, η αντίληψη ότι η Οθωμανική ε, παρακμή ήταν κάτι το αναπόφευκτο, όλα αυτά, καθώς η αντίληψη ότι η Τουρκία θα ήταν πάντα στην περιφέρεια της Ευρώπης χωρίς καμία άλλη αναρκτική λύση από την ένταξη στην Ένωση, όλα αυτά έχουν αλλάξει. Ορισμένοι λένε ότι η Τουρκία μπόρεσε να ξεπεράσει το πρότυπο ενός μη θρησκευτικού, εξυγχρονιστικού αλλά και στρατοκρατικού κράτους. Γιατί αυτό το τύπο, αυτός ο τύπος κοινωνίας και κράτους δεν ήταν οικονομικά αποτελεσματικός. Υπάρχει λοιπόν κάποιος εκδημοκρατισμός και η χορήγηση περισσότερων δικαιωμάτων στην, ε, στο Ισλαμικό τμήμα της κοινωνίας ορίζει και τα όρια του εκδημοκρατισμού και τα όρια της δυνατότητας ε, ενοποιητικού ρόλου στην περιοχή. Ήδη αναφέρθηκε ότι η Τουρκία δεν έθεσε προϋποθέσεις. και ότι έχει ισχυρή πολιτιστική μονόπλευρη αντιμετώπιση, εξωτερική πολιτική. Για παράδειγμα, στα Βαλκάνια η Τουρκία υποστήριξε τους μουσουλμάνους, τα μουσουλμικά κράτη. Το ανέφερε ο Ερντογάν στην ομιλία του για τα Βαλκάνια, όπου παρουσίασε την κυβέρνησή του ως ε, το σωτήρα των καταπιεσμένων μουσουλμάνων. Αλλά μέχρι την Αραβική Άνοιξη η Τουρκία είχε πιο ισορροπημένη άποψη έναντι όλων των διαφόρων ομάδων και κρατών στην περιοχή. Για παράδειγμα τους ε, Σουνίτες, τους Ιήτες, τους Αλεβί, ακόμη και τους Κούρδους στο Ιράκ. Μέχρι στιγμής η Τουρκία είχε μία αντίληψη για μια γενική μουσουλμανική ταυτότητα, όχι συγκεκριμένα δόγματα και ε, μειονότητες. Δηλαδή η Τουρκία θεωρεί τον εαυτό της ως μια μουσουλμανική κοινωνία που βεβαίως είχε διάφορες πλευρές αλλά που είχε ταπεινωθεί από τους Ευρωπαίους απεικιοκράτες και έπρεπε να επανακτήσει την αξιοπρέπειά της. Μετά την Αραβική, Αραβική Άνοιξη η Τουρκία ερμήνευσε τις εξελίξεις με βάση τη δική της εσωτερική ε, εξέλιξη και ε, ενίσχυσε τις νέες δυνάμεις στην ε, την Ισία και την Αίγυπτο. Όμως όταν στη Συρία η κατάσταση βγήκε εκτός κινδύνου και το Ιράν και το Ιράκ ε, ανοιχτά υποστήριξαν το καθεστώς στη Δαμασκό, η Τουρκία ενίσχυσε περισσότερο του Σούνι μαζί με το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία. Οπότε οι σχέσεις με το Ιράν και με την ε, συντηρική κυβέρνηση του Ιράκ επιδεινώθηκαν. Αυτή η αλλαγή έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Συρία, οπωσδήποτε. Βλέπουμε λοιπόν πώς οθήθηκε σε μια ακραία σουνητική θέση η Τουρκία. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τις βασικές θέσεις ε, του ΑΚΠ και του Υπουργού Εξωτερικών που από την αρχή είχαν μια τέτοια θεώρηση της εξωτερικής τους πολιτικής. Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα η Τουρκία κατηγορείται και επικρίνεται όχι μόνο γιατί υποστήριξε τους αδελφούς μουσουλμάνους αλλά διότι δεν έχει, ε, δεν έχει σχέσεις με άλλα τμήματα της Συριακής κοινωνίας όπως τους Δρούζους και τους Κούρδους. Κατηγορείται επίσης ότι έχει προειδοποιήσει τους Σύρους ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί αυτόνομη κουρδική επικράτεια στη Βόρεια Συρία. Άρα θεωρείται ότι οι Τούρκοι ενισχύουν τους Σουνίτες και ότι δεν ενισχύουν και προσπαθούν να περιθεριοποιήσουν τους Κούρδους και τους ε, Δρούζους. Μόνο εάν η Τουρκία καταφέρει να καταλάβει ότι η πολιτική της δεν πρέπει να ευνοεί και να θέτει σε δυσμενή θέση διάφορα τμήματα της ίδιας της δικής της κοινωνίας όταν δημιουργήσει μια έννοια υπηκότητας που δεν θα κάνει διακρίσεις κατά των πολιτών της τότε μόνο θα μπορέσει να παίξει θετικό ρόλο και στην εξωτερική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να, να δώσω το λόγο σε κάποιους βεβαίως ε, αλλά πρέπει να έχουμε και χρόνο για τους βουλευτές μας να κάνουμε ερωτήσεις και, και να έχουμε και απαντήσεις γιατί στις 11 πρέπει να τελειώσουμε να δώσω λοιπόν το λόγο πρώτα απ' όλα στον κύριο Ντανζάου Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους θαυμάσιες, ε, πολύ χρήσιμες Σχόλιο. Συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Γκιοεξέλ. Πολύ σημαντικά. Η επιρροή της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής στην γειτονία της εκφράζεται πολύ λιγότερο και τα αποτελέσματα είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματικά από την διπλωματία ή τις πολιτικές πρωτοβουλίες ή την ε, επιδίωξη δημιουργίας μιας πολιτιστικής ταυτότητας, πολύ λιγότερο από αυτά και πολύ περισσότερο από αυτά που είδαμε στην δεκαετία του 90 μετά την κατάρρευση της Ιουκοσλαβίας. Όλα αυτά έδωσαν πολύ λιγότερα αποτελέσματα από την ε, οικονομική επίδραση της Τουρκίας τώρα. Κυρίως οικονομικά δρούν οι Τούρκοι και η πολιτική είναι παράρτημα. Στη δεκαετία η εξωτερική πολιτική ε, προσπάθησε να επεκταθεί πολύ στην ε, Κεντρική Ασία, τις πρώην ε, Σοβιετικές Δημοκρατίες. Αυτά απέτυχαν. Αλλά τώρα μπορεί να επανέλθει αυτή η προσπάθεια μέσω μιας πιο κοινωνικής και οικονομικής κατεύθυνσης. Χρόνια μας έλεγαν ότι ο κύριος Νταβούτογλου έχει τρομερή στρατηγική σκέψη και οι προσπάθειές του να μην υπάρχουν καθόλου συγκρούσεις με τους γείτονές του, αυτή η πολιτική ειρήνευση τη εξωτερική πολιτική τη Τουρκία, ότι η Τουρκία θα ήταν γέφυρα διαμεσολαβητή, αυτή η πολιτική ε, αντικειμενικά απέτυχε. Οι συγκρούσει ε, έχουν ξεσπάσει παντού γύρω από την Τουρκία, αναθερμαίνονται ακόμη και σε περιοχέ όπου δεν υπάρχουν πραγματικέ συγκρούσει. Πώ λοιπόν το ΑΚΠ προσπαθεί να βιώσει και να μετατρέψει αυτή την αποτυχία ούτως ώστε να υπάρξει μια νέα όθηση. Κατά τη γνώμη αυτή η νέα όθηση είναι ότι αντί για γέφυρα και μεσολαβητής η τουρκική εξωτερική πολιτική γίνεται ενεργός παράγων που παίρνει θέση υπέρ του ενός ή του άλλου ίσως όχι να παίρνει θέση υπέρ αυτού που θα θέλαμε είτε στην Ισραηλινή Αραβική διένεξη, είτε στη σχέση με το Ιράν για τα πυρηνικά θέματα, είτε για τα αφρικανικά θέματα όπως τη Σομαλία, όπου οι σχέσεις με τις Ισλαμιστικές ε, ομάδες είναι τουλάχιστον ε, συζητήσιμες. Θα ήθελα τις αντιδράσεις σας από αυτού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντανζόν είναι πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην Άννα Γκόμες, συντονίστρια των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ε, παρουσιάσεις που ήταν ε, συναρπαστικές και τις συγκεκριμένες προτάσεις ε, της κυρίας Γκέξελ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Τι θεωρείτε ότι είναι ο κύριος παράγοντας ε, της ε, στασιμότητας ε, των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας οφείλεται στην επικριτική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό ή έχει σχέση με την προσέγγιση της Τουρκίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης ε, βρήκα συναρπαστικό αυτό το οποίο είπατε για τα όρια του τουρκικού μοντέλου στην Αραβική Άνοιξη ε, που σχετίζονται με το ότι υπάρχουν περισσότεροι δημοσιογράφοι λεξιμένοι στην Τουρκία από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και αυτό από μόνο του βεβαίως είναι προβληματικό. Αλλά πώς βλέπετε παραδείγματο χάρη την τοποθέτηση της Τουρκίας σε σχέση με την Αίγυπτο. Το Κάιρο πράγματι είχε πολύ μεγάλη σημασία, το τονίσατε, αλλά ε, τονίσατε και τις αντιφάσεις. Και τέλος ε, το Ιράν. Υπήρχαν παραδείγματο χάρη προσπάθειες ε, μαζί με τη Βραζιλία για να αναλάβετε μία πρωτοβουλία για το Ιράν. Πώς βλέπετε λοιπόν το θέμα με τη Σύρια τα ζητήματα μεταξύ Σουνιτών και Σιητών και την ε, σχέσεις με το Ιράν και το διμερές ε, πλαίσιο σε σχέση με τις παγκόσμιες προκλήσεις του Ιράν. Ευχαριστώ, ο κύριος Νταφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά, χαρά μου να Ακούω και πανεπιστημιακού αλλά μιλάνε. καλό είναι το το αυτό. Να ακούμε ανθρώπους που τα ξέρουν τα, τα παράγματα, ακαδημαϊκούς. Έχω ένα σχόλιο που θα μπορούσε να είναι και ερώτηση. Η ερώτηση είναι, θα έπρεπε θα πρέπει ε, ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός Ερντογάν να μετασχηματιστεί σε πρόεδρο Ερντογάν. Ποιες είναι οι πιθανές συνέπειες για την ε, τουρκική εξωτερική πολιτική. Βέβαιως, κασίες κάνουμε γιατί ε, υπάρχουν και οι προεδρικές εκλογές στην ε, Κύπρο την Άνοιξη. Αν ο νέος πρόεδρος της Κύπρου είναι ο κύριος Αναστασιάδης και ζητήσει η Κυπριακή Δημοκρατία να ενταχθεί στην ε, συνεργασία για την ειρήνη του ΝΑΤΟ τι θα γίνει. Και αυτό το ρωτάω γιατί στο τέλος του επόμενου έτους θα έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα αφορά την πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Και κύριος Ερδογάν ε, βεβαίως ε, θέλει πάρα πολύ να εμφανιστεί σε κάποια τέτοια οικογενειακή φωτογραφία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και βέβαια σε αυτό το ερώτημα αφορά και το Κοινοβούλιο. Εμείς θεωρούμε πως θέλουμε να, να ασκήσουμε πίεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να οικοδομήσει γέφυρες ή να ξαναοικοδομήσει ε, μια γέφυρα με την Άγκυρα η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε κακή κατάσταση. Ευχαριστώ. Κύριος, η κυρία. Κυρία Κρόμπερ. Ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσεις. Ο κύριος Ζόιφερτ ε, ανέφερε την στρατιωτικοποίηση της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής απέναντι στη Συρία και την Κύπρο και την Τεχεράνη. Από την άλλη, η Κύπρος έχει παίξει ενδιαφέροντα ρόλο. Και έχει παίξει ενδιαφέροντα ρόλο σε σχέση με το Ιράν και τη... σε συνεργασία με τη Βραζιλία. Πώς βλέπετε λοιπόν τις μακροπρόθεσμες ανησυχίες ασφαλείας και ποιες ε, ασφαλείες, ε, απειλές θεωρεί ότι έχει η τουρκική πολιτική ασφαλείας. Και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις ε, στο Ιράν λόγω των πυρηνικών και είμαι σίγουροι πως αυτές επηρεάζουν και την οικονομία της ε, Τουρκίας. Πώς βλέπετε λοιπόν το ζήτημα των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις ε, σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κυρία Κρόνμπεργκ, είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας για το Ιράν. Ο κύριος Τάνοκ, συντονιστής των Ευρωπαίων Συντηρητικών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να επαναλάβω τα λόγια του Άντριου Νταφ. Ήταν πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα και λόγια ανάλυση του πώς ε, βλέπουν ε, αυτοί οι οποίοι παρακολουθούν την Τουρκία την ε, διαδικασία αυτή αντιμετώπισης ε, των διλημάτων από μια ήπια Ισλαμιστική κυβέρνηση. Και βεβαίω την ανάδυση μίας ε, σουνητική ε, περιφερειακής δύναμης όπως είπε η κυρία Γκόμε. Νομίζω ειδικά οι κυρίες του και Γκουξέλ τα ανέπτυξαν πολύ καλά. Να σας πω τώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα μια ερώτηση. Χτες Ήμουν σε ένα συνέδριο για τα βασανιστήρια και μας είπε κάποιος από το Ηνωμένο Βασίλειο πως καταφτάνουν ακόμα Κούρδοι που έχουν βασανιστεί στην Τουρκία. Ισχύει αυτό και αν ναι γιατί σε μια χώρα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το άλλο το οποίο δεν αναφέρθηκε είναι ο ρόλος Τουρκίας στην Κεντρική Ασία. Όταν συναντάω εγώ ηγέτες από χώρες ε, τουρκογενείς ε, πάντα είναι κάπως επιφυλακτικοί όσον αφορά τις φιλοδοξίες της ε, Τουρκίας στην περιοχή. Επίσης αναφέρατε ε, το ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΑΣΕ. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα σε σχέση με την με το ότι βεβαίω η Ισλαμική διάσκεψη στην οποία είστε μέλο ψηφίζει συνήθω συντεταγμένη για ζητήματα που αφορούν το Ισραήλ ε, κτλ. Και βεβαίως ε, πότε θα ανοίξετε τα σύνορά σας ε, με την Αρμενία. Αναφέρατε πως η αλληλεγγύη με το Αζερβαϊτζάν φτάνει σε σημεία μη κριτική της αζερικής κυβέρνησης. Και εδώ πέρα θα υπάρξει βεβαίως μια μη ταύτιση συμφερόντων ε, όσον αφορά τον Αγκόνο Καρμπάχ. γιατί την δε Κύπρο πότε θα σκεφτείτε κάποια λύση για τα Βαρόσα και την Αμόχωστο ως, μέτρα, ε, ε, ως ένα μέτρο οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Η πόλη είναι μια πόλη φάντασμα και τα κτίρια καταραίων. Ντροπή και, και σπατάλη επίσης. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν θα μπορούσε να γίνει κάτι όσον αφορά την Αμόχωστο και τα Βαρόσα. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλες ε, παρεμβάσεις. Τότε και εγώ που είμαι η συγγήτρια έχω κάποιες ερωτήσεις. Τι θέλουμε τι θέλουμε να κάνει η Τουρκία στην εξωτερική πολιτική. Θέλουμε να αποτελέσει μια γέφυρα προς τη Μέση Ανατολή το πρώτο είναι αυτό. Και αυτό το οποίο είπατε είναι πως η Τουρκία στην αρχή θεωρήθηκε υπόδειγμα στη Μέση Ανατολή. Αλλά βεβαίω δεν μπορούσε να συνεχιστεί κάτι τέτοιο. Μήπως ο λόγος είναι πως, αν δούμε την Αίγυπτο, πως οι αδελφοί μουσουλμάνοι είναι πιο συντηρητική από το ΑΚΠ. Δεν είναι πλέον κοσμική, ενώ το ΑΚΠ οφείλει να είναι κοσμικό. Και επίσης αναφερθήκατε όλοι στα εσωτερικά προβλήματα. Μία από τις βασικές δυσκολίες στην Τουρκία όπως ε, είναι το ότι δεν έχει πραγματική αντιπολίτευση. Γιατί αν είναι να λύσουμε το κουρδικό. Χρειάζεται το CHP και το MHP που ποτέ βεβαίως δεν θα συνεργαστούν. Ούτε η δικαιοσύνη βεβαίως. Και μετά ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χτες είδαμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης με ένα πακέτο το οποίο μας παρουσίασε και το ενδιαφέρον είναι πως ακόμα και όταν δεν ανοίγουν τα κεφάλαια έχει κάποια κάποια άτυπα μέτρα για τις μεταρρυθμίσεις την ε, δικαιοσύνη. Ποιε είναι λοιπόν οι δυνατότητε να γίνει κάτι όσον αφορά τη θετική αυτή ατζέντα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ε, πέντε λεπτά στον κάθε προσκεκλημένο μας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την κυρία Γκεξέλ. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω μερικές ε, από τις ερωτήσεις που θεωρώ ότι με αφορούν περισσότερο και φαντάζομαι πως οι συναδελφοί μου θα απαντήσουν τις υπόλοιπες. δεν ξέρω την ε, απάντηση στο ερώτημα για την Αίγυπτο, αλλά να σας δώσω το παράδειγμα της Τινησίας, όπου η κοινωνία των ε, πολιτών και η αντιπολίτευση ήταν απογοητευμένοι για το ότι το ΑΚΠ έχει εμπλακεί στη χώρα μόνο με τους αδελφούς μουσουλμάνους. Χρήματα, εκπαίδευση, επισκέψεις ε, στο κόμμα που έχει ήδη την εξουσία και δεν προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιον πιο δίκαιο ανταγωνισμό. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι προς το συμφέρον του ΑΚΠ. και βεβαίως, εντάξει, δικαίως, αλλά όπως θα έπρεπε και κάποιοι άλλοι φορείς της Τουρκίας να κάνουν κάτι άλλο με άλλους φορείς της Τινησίας για να είναι έτσι κάπως πιο σφαιρική η τουρκική παρουσία στο μέτωπο που υπάρχει δυνατότητα επιρροής. Τώρα για την ήπια αυτή ισχύει. Συμφωνώ με το σχόλιο πως συχνά είναι οι μη κρατικέ ε, πρωτοβουλίες αυτές οι οποίες εμπνέουν έχει επιχειρηματικός τομέας, ε, σύριαλ τηλεοπτικά, ε, πόλεις ζωντανέ όπου μπορούν συντηρητικοί να συνεπάρχουν με φιλελεύθερους. Ε. Αυτά έχουν τονίσει και οι Τούρκοι πανεπιστημιακοί. Και τι μπορεί να κάνει τώρα η Τουρκία Αυτά θα βοηθήσουν και την ε, Τουρκία, δηλαδή η αλληλεπίδραση με τη Μέση Ανατολή όσον αφορά την ε, ποικιλομορφία και τη δημοκρατία στην ε, Τουρκία. Τώρα το ερώτημα για, για το εάν η Τουρκία, το ΑΚΠ ή κάποιες άλλες δυνάμεις είναι πολύ Ισλαμιστικές και δεν θεωρούν την Τουρκία υπόδειγμα. Ναι, και αυτό ισχύει και φαίνεται στις δημοσκοπήσεις όπου η Τουρκία δεν θεωρείται αρκετά θρησκευόμενη. Αλλά ισχύει και το άλλο. Δηλαδή κάποιες από τις απαντήσεις είναι πως η Τουρκία είναι πολύ θρησκευτικό κράτος ε, και βεβαίως και η τουρκική κυβέρνηση προσανατολίζεται προς τα θρησκευόμενα τμήματα του πληθυσμού. και μια επιφύλαξη. Δεν εννοούσα ότι δεν μπορεί να είναι μοντέλο η Τουρκία. Είναι υπόδειγμα, αλλά η ποικιλομορφία της είναι η προσθέμενη αξία. Εάν χάσει αυτή την ποικιλομορφία, αυτό θα έχει αρνητικές ε, συνέπειες ε, για το κατά πόσο μπορεί να είναι υπόδειγμα για χώρες ε, όπου υπάρχει κίνδυνος για τον πλουραλισμό. Δύο ερωτήσεις τώρα που είναι, με αφορούν άμεσα. Η Αρμενία. Αυτό είναι άλλο θέμα. Υπό την έννοια πως ε, το ζήτημα των συνόρων είναι ζήτημα στρατηγικών συμφερόντων της ε, Τουρκίας. Δεν νομίζω πως είναι απλά προέκταση ε, του, του να μην θυγεί η αζερική κυβέρνηση. Είναι θέμα και της τουρκικής ε, κοινή γνώμης που δεν θέλει να υποχωρήσουμε όσον αφορά τους Αζέρους που θεωρούν θεωρούν θύματα. Στην Τουρκία λοιπόν πραγματικά θεωρούν πως αυτή, από τη στιγμή που θα ανοίξουν τα σύνορα με την Αρμενία δεν υπάρχει πλέον κανένα κίνητρο για να διαπραγματευτεί η Αρμενία με το Αζερβαϊτζάν για το Καραμπάχ. Οπότε είναι πολύ πλευρό το ζήτημα, δεν αφορά μόνο την αλληλεγγύη. Τα ωφέλη του ανοίγματο των συνόρων ε, δεν είναι τόσο μεγάλα σε σχέση με τις αρνητικές συνέπειες που υπάρχουν και από πλευράς ενεργειακής ασφαλείας και μεγάλων επενδύσεων ε, μεταξύ Τουρκίας και Αζερβαϊτζάν. Οπότε καμία κυβέρνηση τουρκική δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι και ζήτημα εθνικιστικό και άρα είναι μια στιγμή δύσκολη για να θίξει τους εθνικιστές ε, η Τουρκία. Δηλαδή άμα είναι να θίξει τους εθνικιστές μπορεί να το κάνει για το κουρδικό που μας καίει αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι λίγο περίπλοκη η κατάσταση στον Καύκασο. Οπότε δεν είναι μόνο ζήτημα Αζερβαϊτζάν. Πρέπει να τελειώσετε, λέει η πρόεδρος. Ωραία, τελείωσα. Ο κύριος Ζόιφερτ. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με την ερώτηση του κύριου Νταουζό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η οικονομία διαρματίζει πολύ σημαντικό ρόλο και όταν ε, και μίλησα για την αύξηση του εμπορίου και της ε, σχέσεις ε, μεταξύ των ε, εμπορευμένων. Η, η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα στην περιοχή που ενδιαφέρεται στην περαιτέρω ανάπτυξη των ε, γειτονικών σχέσεων από οικονομική σκοπιάς να είναι λοιπόν μια προσοδοφόρος σχέση αυτή με τα γειτονικά κράτη. Οι άλλες χώρες περιοχές είναι πετρελοπαραγωγή, παραγωγή φυσικού αερίου και έχουν σε σχέση με την ε, Ευρώπη. Για την ε, Τουρκία λοιπόν έχει μεγάλη σημασία να δημιουργήσει οικονομικούς, πολιτικούς και εμπορικούς δεσμούς με την περιοχή. Θα πρέπει λοιπόν να βασιστούμε στην Τουρκία όταν εμείς ως Ευρωπαίοι θέλουμε να έχουμε λόγο στην περιοχή αυτή. Δεύτερον, να αναφερθώ στα όσα είπε η κυρία Ρόν και ο κύριος Νταφ. τι θα γίνει αν ε, γίνει πρόεδρος ο κύριος Έρδογαν. Η κυρία Βούιτεν ε, είπε ότι έχουμε κάποια κινήματα προοδευτικά και τι γίνεται τώρα. Η αντιπολίτευση δεν είναι σε θέση να ε, παρεμποδίσει τον Έρδογαν να εκλεγεί πρόεδρος και δεν μπορεί να κάνει τίποτα από την άλλη μεριά για να προωθήσει τη δημοκρατία. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πολιτευσή δρά προ την κατεύθυνση αυτή. Ακούσαμε ότι 60 βουλευτέ του Κοινοβουλίου συμφώνησαν με την πολιτική του ΑΚΠ για να ε, αρθεί η ασυλία ε, βουλευτών. Είδαμε λοιπόν ότι αυτό το συντηρητικό κόμμα είναι το κόμμα το οποίο ε, στηρίζεται από το μεγαλύτερο σώμα της κοινωνίας. Θα πρέπει λοιπόν να εμπιστευτούμε και να ενθαρρύνουμε αυτή την πολιτική διαφοροποίηση σε αυτό το πολιτικό φάσμα. Χρειάζεται λοιπόν να στηρίζουμε αυτού του είδους τις διαφοροποίησεις και να πάψουμε, πάψει να υπάρχει αυτή η απόλυτη αντιπολίτευση και αντίθεση με την Τουρκία, διότι, την πολιτική Τουρκία, διότι αυτό ε, αναπαράγει μια εσφαλμένη και επικίνδυνη πολιτική. Ένα άλλο ζήτημα ήταν αυτό που είπε η κυρία Γκόμες, ε, για να πω κάτι προκλητικό. Ζήτησε Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα για την ένταξη. Είναι η πολιτική της κυβέρνησης, είναι η Κύπρος. Ακούγεται παράδοξα, αλλά όταν μιλάμε τόσο πολύ για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζουμε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία. Ίσως θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με το ζήτημα το κατά πόσον θέλουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία για λόγους ε, αναπτυξιακούς, για λόγους ασφάλειας και για ένταξη των ε, μεταναστών. Για όλους τους λόγους λοιπόν θα πρέπει να οικοδομήσουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία και να λάβουμε υπόψη ότι η Τουρκία σήμερα δεν ε, επιθυμεί τόσο πολύ να καταστεί πάση θυσία μέλος. Χρειάζεται λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα πιο ήπια, πιο ήρεμα. Όταν λοιπόν η Τουρκία φτάσει στο σημείο να λάβει την απόφαση, ενδεχομένω και να πει όχι. Για μας σημασία έχει να αποκτήσουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία και να ξεφύγουμε αυτόν τον πανικό που επικρατεί. Και τέλος ε, Κύπρος δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο συμβασμό τη Τουρκία στο κυπριακό ζήτημα και εδώ δεν έχω κάποια απάντηση. Ω εκ τούτου πιστεύω ότι η Τουρκία στο τέλο δεν θα καταστεί μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η διαδικασία διαπραγμάτευση δεν θα προχωρήσει εφόσον η Τουρκία θέλει να ε, καταστεί περιφερειακή δύναμη τώρα η στρατηγική, η στρατιωτική πάντα μιλούσαν για τη στρατηγική σημασία της Κύπρου. Αλλά σήμερα με τη νέα κατάσταση που επικρατεί με την Κύπρο, το Ισραήλ, την Ελλάδα και με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή η Κύπρος είναι ένας ε, στρατηγικός παράγοντας ε, Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο επί του τελευταίου. Ναι, ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με το ερώτημα της κυρίας Γκόμες για το γιατί έχουμε στασιμότητα. Διάφοροι παράγοντες ε, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Τουρκία. Είναι προφανής ε, το Κυπριακό που μπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις. Επιπλέον έχουμε αντιφατικά μηνύματα, ειδικά από το 2005 και μετά για το εάν η Τουρκία θα ενταχθεί ή όχι. Το εάν θα είναι κάποιος προνομιούχος εταίρος και από τις πρωτεύουσες, ε, τη Γαλλία, η Γερμανία, ε, Σαρκοζή που, ε, και το φαινόμενο Σαρκοζή που εξακολουθεί να υφίσταται και όλα αυτά έπαιξαν μεγάλο ρόλο. Η αίσθηση στην Τουρκία είναι πως η Τουρκία δεν έχει προοπτική ένταξης. Και αυτός είναι παράγων βεβαίως ε, στασιμότητας, αλλά αυτό το οποίο επίσης συμβαίνει είναι πως ε, η δημοκρατία αρχίζει να σκοντάφτει, μετά έχουμε κάποιες επιλογές στην εξωτερική πολιτική που είναι ad hoc και όχι τόσο συστηματικές και υπάρχει μια μεταβολή μετά και στην τουρκική πολιτική και κοινωνία. Και αυτό που με ανησυχεί είναι πως εάν συνεχιστεί κάτι τέτοιο τότε κάποιες από αυτές τις αλλαγές θα γίνουν μόνιμες ή έτσι πιο εδρεωμένες Σε αφορά δηλαδή τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό που υπήρχε στην ε, τουρκική κοινωνία και στην ε, τουρκική νεολαία παραδείγματος παρά τα όσα υπήρχαν με εθνικισμό κτλ. Αυτό μου ανισχύει. Επίσης για το Ιράν αυτό το οποίο συνέβη και το λέω και αυτό στα μαθήματά μου όταν ε, ήταν παρούσες η ΙΠΑ στο Ιράκ η Τουρκία έκανε μια εξωτερική πολιτική στη σκιά των, των ΙΠΑ και θεωρούσε πως η σκιά αυτή ήταν δικιά της και όταν έφυγαν οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, έμεινε η σκιά του Ιράν γι' αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή έναν ανταγωνισμό δυνάμεων στην περιοχή και μάλιστα όταν προσπαθεί κανείς να αναλύσει τις επιλογές εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή. Πέρα από την ιδεολογία και τον Ισλαμισμό, καλύτερο είναι να το δούμε ως ένα παιχνίδι ισχύω, κυρίως με το Ιράν ως ανταγωνιστή. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα του κυρίου Νταφ για το τι θα γίνει αν ο Ερντογάν γίνει πρόεδρος. Εδώ πέρα βεβαίως δικασίες θα κάνω. Πρώτα απ' όλα ναι, φαίνεται πως θα γίνει ε, πρόεδρος ε, προφανώς δεν μπορούν να αλλάξουν το, το σύνταγμα από μόνοι τους. Είναι προφανές πως όλα τα άλλα κόμματα είναι εναντίον. Το BDP μπορεί να μην είναι εναντίον, αλλά εξαρτάται από το τι θα λάβει ως αντάλλαγμα. Και δεν ξέρω αν θέλει να του δώσει αντάλλαγμα το Ερντογάν. Επίσης, υπάρχει η ε, πιθανότητα, η οποία υφίσταται και, και οφείλω να το πω, το ανέφερε και ο κύριος Ζόιφερτ. Ναι, ανταγωνισμού όχι βεβαίως από το Τσέχαπε. Α, μιλάμε για την περίπτωση που γίνει δημοψήφισμα και εγκριθεί κτλ. Και, και βεβαίως ε, τίθεται το ζήτημα μετά για το εάν θα υπάρξει κάποιος ε, ανθυποψήφιος από αυτό το κόμμα. Είναι πιθανόν. Αλλά αν δεν γίνουν αυτά και γίνει πρόεδρος ο Ερντογάν, τότε ε, εγώ θα ήθελα να είμαι αισιόδοξη και να πω πως ε, θα μπορούσε να είναι πιο τολμηρός ε, και λιγότερο εθνικής, γιατί δεν θα χρειαζόταν, δεν θα χρειάζεται πλέον να είναι. Οπότε έτσι αν πάνε οι κυπριακές εκλογές όπως λέτε ότι θα πάνε, ίσως έχουμε μια ευκαιρία. Ε, ίσως λοιπόν ε, έχουμε και μια ευκαιρία μετά και στο κουρδικό μέτωπο. Και τέλος για τα σχόλια του κυρίου Τάνοκ για τα βασανιστήρια. Υπάρχει και η τελευταία έκθεση του Χάμαρμπεργκ από το Συμβούλιο της Ευρώπης που λέει πως μειώνονται τα βασανιστήρια. Δεν είναι συστηματικά όπως ήταν στη δεκαετία του 90 αλλά ακούμε περιπτώσεις ε, κυρίως ε, ατιμορρησίας σε μέρη της δικαιοσύνης και της αστυνομίας. Για την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν, κοιτάξτε, η συμφωνία μας η τελευταία με το Αζερβαϊτζάν μπορεί να ακούγεται καλή, αλλά αναφέραμε και τα της Αρμενίας, οπότε εκεί πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Τώρα για τα δικά σας σχόλια για το τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό το οποίο παρατηρώ είναι η τάση να αποσυνδέονται να αποσυνδέεται η δεξιακή προοπτική και να μιλάμε μόνο για μια συνεργασία χωριστή κάτι το οποίο εγώ θεωρώ πως είναι προβληματικό επίσης ε, η δικαιοσύνη είναι πραγματικά προβληματικός τομέας μεταρρύθμισης είναι ο βασικός τομέας διαφωνίας δηλαδή ποια είναι τα προβλήματα της ε, δικαιοσύνης είναι το υπερβολικό βάρος, ε, ενώ βεβαίως είναι ταυτόχρονα και ανεξάρτητη η δικαιοσύνη και υπάρχει και ζήτημα αμεροληψίας. Και βέβαια η κυβέρνηση ασχολείται μόνο με το ζήτημα του υπερβολικού βάρους ε, εργασίας. Το ΤΣΕΧΑΠΕ τώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση μετασχηματισμού και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανταγωνιστική πολιτική εντός της Τουρκίας. Γι' αυτό ακριβώς ε, κινδυνεύει θα έλεγα η δημοκρατία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Πρέπει να συνοψίσουμε αλλά και ο κύριος ε, Ριπέρτο, ο πρέσβης πρέπει να λάβει το λόγο και προτείνω να συνοψίσετε εσείς. Ευχαριστώ. Δεν είμαι θα ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα πάνω στα ζητήματα που θίξατε. Τώρα, ποιοι είναι οι λόγοι για την ε, στασιμότητα. Ένα τμήμα τη ευθύνη το φέρουν τα κράτη-μέλη και στην Τουρκία σε ό,τι φορά την διαπραγμάτευση επί των κεφαλαίων. όπω γνωρίζετε πολύ καλά. Πολλά κεφάλαια έχουν μπλοκαριστεί από το Συμβούλιο ή από τα κράτη-μέλη. Και de facto τα τρία εναπομείνοντα έχουν ε, λίγο πολύ παγώσει λόγω Τουρκίας και ελπίζουμε το σύντομα, πολύ σύντομα, χάρη ε, ε, στις εξελίξεις ε, που μπορούν να προέρθουν από την Γαλλία και την Τουρκία θα μπορούσαν να προοδεύσουμε. Ας είμαστε ξεκάθαροι όμως να πούμε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα από πλευρά της Τουρκίας, να βλέπουμε την κρίση στην Ευρωζώνη, την οικονομική κρίση κλπ. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα εδώ και αν και ο πλευράς ε, επιχειρηματιών ε, αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν ε, προβλήματα, έχουν υπάρξει, έχει, έχουν, έχει υπάρξει πρόοδο σε ό,τι φορά το οικονομικό κομμάτι. Το θέμα της Ισλαμοφοβίας δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Δεν υπάρχει Μάλλον είναι δεχόμενο να προκύψει κάτι τέτοιο και ε, φυσικά μπορείτε να αναρωτηθείτε για το 100% ε, του κεκτημένου να έχει ολοκληρωθεί πριν από την πραγματική, μετά από την ουσιαστική πρόσβαση, ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό. Να πω κάτι για το τουρκικό μοντέλο. Έχει μεγάλη σημασία για ορισμένε χώρε ε, όπου ε, έχουμε αναδυόμενη δημοκρατία ε, ότι οι εξελίξη στην Τουρκία οδήγησαν στο να υπάρξει ένας εκδημοκρατισμός. Αυτό είναι σημαντικό για την Τουρκία, για την, Ισία. Τώρα για το, προ... για το κατά πόσο είναι ελκυστικό αυτό το μοντέλο, αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα εάν του ρωτάτε τον κόσμο εάν ε, θεωρούν την Τουρκία δημοκρατία και απαντούν ναι, τότε φυσικά θέλουν και αυτοί να έχουν ένα παρόμοιο καθεστώς. Τώρα ας λάβουμε υπόψη ότι αυτό το οποίο συνέβησαν στη Γάζα είναι πολύ σημαντικά και η Τουρκία έχει γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος εταίρος της ε, Αιγύπτου μετά την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από την, Ιαπωνία, μετά από την Κίνα. Αυτό έχει σημασία. Πάντως η Αίγυπτος παραμένει η, σημαντική δύναμη στην περιοχή. Αυτό το σκέφτεται πολύ καλά η Τουρκία. Εμείς πάντως γνωρίζουμε τις εκθέσεις που έχουν συνταχθεί και βρισκόμαστε σε συνεργασία με τα ΙΠΕΞ για τις συνθήκες κράτησης και της ατιμορρησίας. Αυτά τα πιστεύω στην την ε, περίοδο της ε, απεργίας ε, πείνας κατέδειξε ότι δυστυχώς το πρόβλημα παραμένει και η κυβέρνηση έχει λάβει κάποια ε, στεναρά μέτρα σε ό,τι αφορά την ε, θέση των Κούρδων, Κούρδων θα πρέπει να τονίσουμε κάποια πρόοδο που έχει, επιτευχθεί. Ελπίζουμε η κυβέρνηση να ε, θελήσει να διαπραγματευτεί. Και κάτι ακόμα. εν διαδικασία περί συντάγματος. Θα πρέπει να ε, ακούσουμε τα μέλη της Επιτροπής. Ε, θα συνεχίζουν λοιπόν όλα τα μέρη να συνεργάζονται. Όταν το ΣΥΑ είπε ότι θέλουμε 10 μέρες ε, για να το σκεφτούμε και υπόθηκε εντάξει. Όταν οι ηγέτες του PTP αποφάσισαν να προχωρήσουν σε απεργία πείνας, ε, είπαν ότι ναι, εμείς ως Επιτροπή θα περιμένουμε να επανέλθουν τα μέλη του PTP. Αυτό είναι το πνεύμα. Δεν βλέπω λοιπόν πως ο Πρωθυπουργό ακόμα και αν το επιθυμεί μπορεί να διακόψει αυτή την διαδικασία. Δεν έχουν, δεν έχουν πεντευθεί ιδιαίτερα θετικά, θετικές εξελίξεις, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι ο Πρωθυπουργό ε, θα πρέπει να ε, συνεχίσει προσπάθεια προσπάθειές Τώρα, αν ε, ο Πρωθυπουργό πάρει την θέση του Προέδρου και τι είδους προεδρικό σύστημα θα υπάρχει, αμερικανικό, γαλλικό κλπ. Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Πρέπει να όμως να διατρήσουμε τον Πρωθυπουργό Εντοργάν ε, στο πλαίσιο της ε, συνεννόησης για τη διαδικασία που έχει ξεκινήσει μου. Θα τα αναγνώσετε στην προσεχή έκθεση. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που μας δώσατε νέες φρέσκες πληροφορίες αλλά υπάρχει και κάτι το οποίο θα ήθελα να δω να γίνεται. Αυτό που είπε ο πρέσβης ότι χρειάζεται να ε, αναμειχθούν, να εμπλακούν ε, οι Τούρκοι πολιτικοί, αλλά και περισσότερο παραποτέ θα πρέπει να εμπλακούν και να συμμετέχουν τα κράτη-μέλη. Γιατί αν θέλουμε η Τουρκία να δημιουργήσει ένα ρόλο, τότε η Τουρκία θα πρέπει να είναι ένα ε, υπόδειγμα προτύπου και να πληρεί τα πολιτικά κριτήρια. αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το κράτος να έχει μια ε, ισορροπημένη δημοκρατία αφενός, αλλά αυτό οδηγεί σε υπευθυνότητα της, ε, την αντιπολίτευση, διότι αυτό το οποίο γίνεται τώρα για την κουρδική, κουρδική ε, αντιπολίτευση είναι καλό αλλά το κράτος χρειάζεται μια ανεξάρτητη και ανεξάρ... ε... δημο... Ε, ανεξάρτητο δημοκρατικό ε. uh, part of a conclusion then I would like to thank everybody σύστημα δικαιοσύνης ε, ανεξάρτητο. Δυστυχώς πρέπει να φύγω τρέχοντας διότι πρέπει να πάω σε επιτροπή για να παρουσιάσω μια έκθεση. Ευχαριστώ.